Ε, señor presidente. Καλημέρα σα, κύριε Επίτροπη. Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ξεκινήσει, θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας και πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα το πρωί είναι η συζήτηση για τρεις πολύ σημαντικές εκθέσεις. Η έκθεση που αφορά την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών είναι η πρώτη. Είναι η έκθεση της κυρίας Τούν und Hohenstein στη συνέχεια που έχουμε την, τα αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς και το Solvit, την έκθεση Solvit. Τρεις εκθέσεις λοιπόν. Θα δώσουμε το λόγο στους εισηγητές. Κάθε εισηγητής θα έχει τέσσερα λεπτά στη διάθεσή του για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Σας παρακαλώ να γνωρίζετε ότι στη συνέχεια οι εισηγητές θα έχουν δύο λεπτά στο τέλος της συζήτησης. Θα έχουν δύο λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντήσουν, να αντιδράσουν και τρία λεπτά για την παρουσίαση. Και τρία λεπτά στην, στο τέλος, τρία και τρία έξι, διότι έχουμε και τον κανονισμό για τις δύο αυτές παρεμβάσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα απ' όλα θα λάβει τον λόγο η κυρία Τούν Χόινστάιν, παρακαλώ, για να παρουσιάσει την έκθεσή της. Έχετε τον λόγο συνάδελφε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα την 19η ε, έκθεση που αφορά τις επιδόσεις ε, για την ενιαία εσωτερική αγορά και τους καταναλωτές που κατατέθηκε τον Ιούλιο Περισσία. Αυτό το έγγραφο